Ε, του, κανονισμού για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ούτω ώστε στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Επίτροπε. Ε, ε, ε τελειώσαμε, ε, ήλπιζα να τελειώσουμε πριν από τις 12, τελειώσαμε έγκαιρα, ευχαριστώ ε, τους πάντες, ε, τους συνεργάτες μας και τους διερμηνείς. Ε, ολοκληρώσαμε την διαδικασία και ε, θα συνεχίσουμε από ε, τις 9 μέχρι τις 12, 5η 16 Φεβρουαρίου. Είναι στην διάθεσή μας, θα είναι στη διάθεσή μας τα πρακτικά. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.